ο κύριος Πρόεδρος. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην σημερινή μας ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Το λόγο έχει